Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Γκαρντίνη με θέμα «Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών, ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας». Θα αρχίσουμε την συζήτηση με την εισηγήτρια. Κυρία Γκαρντίνη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν αυτή την εβδομάδα, αυτούς τους μήνες, στην παραγωγή αυτού του εγγράφου που σήμερα ψηφίζουμε στην ε, Ολομέλεια. Εργαστήκαμε, πρέπει να πω, πάρα πολύ καλά και ήταν πράγματι επικοδομητική η συζήτηση. Η πρόταση ψηφίσματος που ψηφίζουμε λοιπόν σήμερα, η έκθεση αυτή, είναι καρπός ε, κοινής δουλειάς και είναι καρπός της συνεισφοράς ε, όλων των πολιτικών δυνάμεων όλου του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι αναπτύχθηκε μια κοινή ευαισθησία πολύ ισχυρή όσον αφορά αυτό το θέμα και πρέπει να θυμηθούμε μάλιστα ότι ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται πράγματι από μια εκθετική αύξηση των καταστροφών. Οι αριθμοί, αν τους δούμε, ε, στην ομοία αλήθεια τους είναι πολύ ευγλωτοί. Ο αριθμός των καταστροφών στον κόσμο έχει πενταπλασιαστεί. Αν σκεφτούμε ότι το 75, το 1975 καταγράφτηκαν 78 ε, γεγονότα καταστροφικά, ενώ σήμερα έχουμε σχεδόν 400 τέτοια γεγονότα καταστροφικά το χρόνο. Τα τελευταία 20 χρόνια δυστυχώς τα θύματα αυτών των καταστροφών είναι 90.000 και πάνω από 29 εκατομμύρια άτομα ε, επλήγησαν από τις καταστροφές ενώ οι οικονομικές απώλειες φτάνουν στα 211 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο, φαινόμενα μάλλον τέτοιων διαστάσεων που απαιτείται μια απάντηση ισχυρότερη, απάντηση αποτελεσματικότερη και μια δέσμευση από την πλευρά μας ε, μεγάλη για να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε όλοι στα μάτια μας τις εικόνες του σεισμού της Αιτής, των πλημμυρών στο Πακιστάν, αυτών που συνέβησαν στην Ιαπωνία. Η Ευρώπη ίδια βλέπει στην επικράτειά της κάθε μέρα διάφορες πυρκαγιές, πλημμύρες ε, ας πούμε θυμηθείτε όταν είχαμε το Ισλανδικό ηφαίστειο και το σύννεφο που προκάλεσε η έκρηξή του όλα αυτά μας δείχνουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο που ακολουθεί δύο θεμελιώδεις αρχές που είναι πολικοί μας αστέρες. Η αρχή της αλληλεγγύης είναι η πρώτη η οποία ενισχύεται από τη ρήτρα αλληλεγγύης της συνθήκης της Σαββόνας και η αρχή της επικουρικότητας κινούμεθα επ' αυτών των γραμμών. Η παρέμβαση Ευρωπαϊκή Ενώσεω ήδη κατά το παρελθόν πάντα ήταν γενναιόδορη, ήταν αποτελεσματική. Μαρτυρία αυτού πιστεύω είναι η δουλειά που έκανε επίτροπό μας η κυρία Γεωργίευα. σήμερα χρειαζόμαστε να κάνουμε ποιοτικό άλμα, ένα ποιοτικό άλμα που είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για να περάσουμε από μία απάντηση ad hoc σε μία απάντηση όπου η αντίδραση προέρχεται από την προληπτική, προληπτικό εντοπισμό των μέσων που διαθέτουν κάτι μέλη και πώς εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό μετά να υπογραμμίσουμε τι πρέπει να κάνουμε το ποιοτικό άλμα. Πώς, πώς πώ πρέπει να διαδίδονται οι πληροφορίε και πώ να πρέπει να ανταπόκριση στι ε, καταστροφέ που χρειάζεται ο έλεγχο, ο συντονισμό, η συνεννόηση. Θεμελιώδη ο ρόλο των υπηρεσιών όπω το GMS και δράτω με τη ευκαιρία για να πω ότι ανησυχούμε για αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά τον προπολογισμό για τις νέες τεχνολογίες που είναι θεμελιώδη σημασία που θέλουμε να πετύχουμε. Έχουμε αναφέρει την, την σημασία που έχει η επικοινωνία με του ε, πολίτε. Είδαμε στην Ιαπωνία, μάθαμε από την Ιαπωνία. Ποτέ δεν αρκετεί αυτή η επικοινωνία, ποτέ δεν αρκεί. Και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την οποία ζητούμε να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατό μια πρόταση σχετικά με την πολιτική προστασία, ε, να μας δώσει μια νομοθετική πρόταση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαρντίνη. Τώρα η Επίτροπος, η κυρία Γεωργίευα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα και είμαι ευγνώμων στην κυρία Γκαρντίνη που προετοίμασε την έκθεση αυτή. Όπως είπε πολύ σωστά, ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχουν οι κλιματικές αλλαγές, το δημογραφικό ζήτημα, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά όπως επίσης και η τρομοκρατία, μας ε, βάζει σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε διαπιστώσει τι ρόλο έχει παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργώντας μεγάλες φιλοδοξίες προκειμένου η αλληλεγγύη να λειτουργεί πραγματικά και για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους πολίτες ολόκληρου του κόσμου. Και εδώ θα αναφερθώ σε πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί εδώ όσον αφορά την καταπολέμηση των ε, πυρκαγιών στα δάση προκειμένου να δημιουργηθούν επιλοτικά προγράμματα όπως ε, το Bad Flood Module, όπως επίσης και για θέματα μεταφοράς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστροφές και πράγματι όλα αυτά μας βοήθησαν πάρα πολύ και στην περίπτωση της κρίσης της Λιβύης. Έτσι λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε όλο και αυξανόμενε ανάγκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τι ευθύνε τη, τι παίρνει πάρα πολύ σοβαρά και γι' αυτό έχουμε προωθήσει μια ανακοίνωση η οποία πλέον παίρνει νομοθετική μορφή και βασίζομαι για να γίνει αυτό όντως πραγματικότητα στη δικιά σας τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανακοίνωση μας αυτή βασίζεται σε τέσσερις αρχές. Η πρώτη είναι ο σεβασμός του κύριου ρόλου των κρατών μελών προκειμένου να ε, διασφαλίζουν την σιγουριά των πολιτών τους, την προστασία των πολιτών τους. Αυτή είναι μια προσέγγιση όπου βάζουμε από κοινού τους πόρους των κρατών μελών προκειμένου να υπάρχει συλλογική δράση. Όταν ε, χρειάζεται την βοήθειά μας ε, μια χώρα εξαιτίας μια φυσικής καταστροφής. Δεύτερον, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να προλαμβάνουμε τους κινδύνους έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να μπορούμε να αντιδράσουμε αποφασιστικά. Αν έχουμε προβλέψει ένα κίνδυνο μπορούμε καλύτερα να τον αντιμετωπίσουμε. Έτσι θέλουμε τα κράτη-μέλη να έχουν σενάρια για τέτοιες περιπτώσεις. Τρίτον, δεν θέλουμε την ad hoc ε, ανταπόκριση όπως είχαμε μέχρι τώρα. Θέλουμε να προβλέπουμε τα προβλήματα. Και τέταρτον, ξέρουμε ότι περνάμε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Γι' αυτό όμως πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε με συνεργασία μεταξύ μας να έχουμε εξοικονομήσεις στα κράτη-μέλη. Σε αυτά βασίζεται λοιπόν η πρότασή μας. Ζητάμε μια ελάχιστη αύξηση που 25-65 εκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως σε αυτή τη βάση δημιουργούμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα αλλά και εξοικονομήσεις στα κράτη-μέλη. Και θα τελειώσω με ένα επικριτικό σημείο. Αυτά όλα τα κάνουμε για τους πολίτες μας. Και πάνω από 90% από τους πολίτες μας θέλουν να δρούμε από κοινού, μαζί, σε συνεργασία, σε περίπτωση τέτοιων καταστροφών. Το οφείλουμε σε αυτούς λοιπόν να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχει προβλεφθεί τώρα εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο κύριος Τόκιος να πάρει το λόγο, ο οποίος δεν φαίνεται ακόμα στην αίθουσα. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Στρίφλερ εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Euh, euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πολλαπλασιασμό των φυσικών καταστροφών των μεγάλων και οι δημοσιονομικέ πιέσει οι τωρινέ έχουν σαν συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει πραγματικά να ενισχύσει τη δυνατότητά τη αντίδραση στι καταστροφέ και να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο του περιορισμένου πόρου που διαθέτει. Μετά από πολλά αιτήματα του Κοινοβουλίου μα, και η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσει νομοθετικού περιεχομένου που θα είναι φιλόδοξε για το τέλο του 2011, ώστε να δημιουργηθεί επιτέλου μια πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη προστασία πολιτική που θα ε, την υποστηρίζουν διάφορα κράτη-μέλη και εθελοντικά θα διαθέτουν διάφορα τμήματα προστασίας πολιτικής προκαθορισμένα και θα είναι έτοιμε οι μονάδε να παρεύουν άμεσα για επιχειρήσει υποστήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών. Ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για την ανακοίνωσή τη όσον αφορά το δημοσιονομικό πολιετέ πλαίσιο 2014-2020. Προβλέπει 455 εκατομμύρια ευρώ, ε, ευρώ για το μέσο τη προστασία των πολιτών και δίνει μεγάλη σημασία στι δράσει προετοιμασία και πρόληψη. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει άοκνα για να υπάρχει ορατότητα των πόρων και πόσο μπορούν να κινητοποιηθούν οι μονάδες επιτόπου μέσω της χρήσης των συμβόλων της Ευρωπαϊκής Ενώσης να προβληθεί αυτή η εικόνα. παρόλληλα με τα εθνικά μπάτζ, να φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πολύ. Τώρα ο κύριο Σταυρακάκη θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κρατήστε το χρόνο, διότι ξέρετε ότι πρέπει να πάμε στι ψηφοφορίε αργότερα. Δεν έχουν πολλά περιθώρια. Ε, κύριο Σταυρακάκη, για ένα λεπτό, από την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και να εκφράσω την ικανοποίησή μου τόσο για την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην πρόληψη και διαχείριση των πυρκαγιών, όσο και για το γεγονό ότι οι κύριε θέσει τη Επιτροπή Ρέτζι ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο ω επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη, τονίζουμε κυρίω το γεγονό ότι η ρήτρα αλληλεγγύη που εισάγεται με το άρθρο 222 τη συνθήκη τη Λισαβόνα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντική βάση για την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη από πλευρά ευρωπαϊκής ένωσης της δράσης των κρατών μελών στον τομέα τη πολιτική προστασία. Τέλο υποθυμίζουμε το ρόλο και την ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών το σημαντικό ρόλο του ευρωπαϊκού ταμείου Περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάγκη αξιοποίηση τη πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε επίπεδο περιφερειών μέσα από τα προγράμματα Περιφερειακή συνεργασία και τέλο ότι οι νησιωτικέ και ορεινέ περιοχέ είναι εξαιρετικά ευάλωτες στι καταστροφέ λόγω τη γεωγραφική του θέση. Κλείνοντα, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία επίτροπο να σχολιάσει το σημείο 7 τη έκθεση για τη συγκρότηση μια δύναμη πολιτική προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Σταυρακάκη. Ήσασταν και σχεδόν ακριβείς στον χρόνο. Εύχομαι και οι υπόλοιποι ομιλητές. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Σίμπερ τώρα. Κύριε Σίμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ε, έκανε το ουσιώδες ε, έφταξε μία συνοπτική έκθεση και αναφέρει τα ουσιώδη στοιχεία τα οποία πιστεύει και έχει ε, ως θέση το Κοινοβούλιο έναντι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα ήταν ε, σωστό να επιβαρύνουμε την έκθεση. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις αρχές. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτό μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε κράτος μέλος. Μία τέτοια φυσική καταστροφή που θα έχει μεγάλη, μεγάλο αντίκτυπο και στις ανθρώπινες ζωές αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Διαπιστώνουμε ότι οι ζημιές αυτές τα τελευταία χρόνια αυξάνονται μαζικά και ότι ο βαθμός ε, σύνδεσης ε, αυξάνεται στην κοινωνία μας και είναι λογική συνέπεια εδώ στην Ευρώπη να πρέπει να καταβάλουμε πιο κοινέ προσπάθειες. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη στην πρότασή τη και το είπε και η Επίτροπος ότι καταρχάς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι πρωταρχικά υπεύθυνα, αλλά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίζει πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο. Και εδώ λοιπόν μία ερώτηση, κυρία Επίτροπε. Είναι λοιπόν προτεραιότητά σας και αρμοδιότητά σας αυτό που συζητάμε. Ωστόσο, ζητάμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να αναλάβει δράση και είπατε εκπρόσωπος. Πολύ ανησυχώ ότι θα προκληθεί ε, μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα ξέρουμε τελικά ποιο είναι ο αρμόδιο και υπεύθυνο. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε εξ αρχή για να μην υπάρχουν επικαλύψει. και σημαντικό είναι να επικεντρώσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και να... Ε, συμφωνήσουμε προκαταρτικά τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μπορούμε να αντιδράσουμε γοργά. Ήμουνα εισηγητή για την οδηγία για τι πλημμύρε. και είδαμε ότι όταν υπάρχει καλή προετοιμασία μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και σε οικονομικό επίπεδο να αποφύγουμε ζημιές. Ελπίζω λοιπόν κυρία Επίτροπε να υποβάλλετε σχετική πρόταση σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίμπερ. Τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών Δημοκρατών ο κύριος Λέντερ για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Και εμείς ε, καλωσορίζουμε την ανακοίνωσή σα για την ε, βελτίωση τη προστασία από καταστροφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουν σε περίπτωση καταστροφών να αντιδράμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Και κυρίω να βοηθάει ο ένα τον άλλον. Κατά το παρελθόν είχαμε μείνει ε, αν θέλετε, πολλέ φορέ άφωνοι και βοήθητοι μπροστά στην τηλεόρασή μα, κοιτώντα τι καταστροφέ σε όλο τον κόσμο και αναρωτιόμασταν γιατί δεν βοηθάμε. Η ανακοίνωσή σας λοιπόν αποτελεί το επόμενο βήμα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, για μια αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τα μέσα που διαθέτουμε στην Ευρώπη. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, πραγματικά. Έχουμε όλα τα μέσα για να απαλύνουμε και να αντιδράσουμε σε καταστροφές. Άρα θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός. Αναφέρθηκε ότι οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να αντικατασταθούν από μια κεντρική διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται συνέργεια όμως. Χρειάζεται γοργή αντίδραση όλων μας. Από κοινού. Αυτό λοιπόν είναι κατεπήγον. Επίσης συμφωνώ ότι όλο και πιο πολύ θα πρέπει να σκεφτόμαστε προληπτικά. Με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να α, δρούμε σωστά, να μην περιμένουμε μέχρι να χτυπήσει η καταστροφή. Σε περίπτωση ενδεχόμενης εξηρασίας, πλημμύρας, πυρκαγιάς και χαίρομαι που από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αντιδράσουμε σε καταστροφές και να οργανώσουμε την αντίδρασή μας όπως και στο εξωτερικό. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Ζέιμπερ. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι αρμοδιότητες. Εσείς είσαστε αρμόδια. Δεν θέλω να υπάρχει μια μεικτή αρμοδιότητα όπου εκ των υστέρων δεν θα ξέρουμε ποιος ήταν αρμόδιος γιατί. Και τελευταίο θεωρώ ότι αυτή η διαρκής ε, ικανότητα αντίδρασης ακόμα και το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, σε αργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ την κυρία Γκουαρτίνη για την καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέινεν. Τώρα εκ μέρου των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριος Σουγγίας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε Γεωργίευα, είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την εισηγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη και τους άλλους και οδησηγητές για την πάρα πολύ κακοφόλα συνεργασία σε πολύ επίκαιρο θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Είμαστε ικανοποιημένοι, όπως έλεγα, για την προσέγγιση που ήταν ισορροπημένη και λογική. Έτσι αντιμετωπίστηκε το θέμα που συμπεριλαμβάνει την αρχή της επικουρικότητας και την ιδέα μιας ρήτρα αλληλεγγύης που θα πρέπει να εμπνέει τις δράσεις των κρατών μελών σε απάντηση που θα δώσουν σε καταστροφές και στην προστασία των πολιτών. Και πιστεύω συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα είναι σχεδιασμένο, προβλέψιμο στα πλαίσια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβόμενο πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και συνεπώς χωρίς να συνεπάγεται τη δημιουργία ενό υπερεθνικού σώματο, που αυτό θα επεκάλυπτε και κόστο και αρμοδιότητε χωρί να έχουμε την εγγύηση τη αποτελεσματική λειτουργία αυτού. Εκφράζω εκτίμηση ιδιαίτερη για την προσοχή που δόθηκε στου εξαίρετα ε, ευάλωτου το, ε, περιοχές όπως είναι νησιά και δίνεται σχέση μεταξύ προετοιμασίας, πρόληψης και απάντησης στις καταστροφές. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αποτελούν μια τριάδα που είναι απαραίτητη. Στέλος, χρειάζεται προσοχή όσον αφορά την ευαισθησία που έδειξαν οι συνάδελφοι όσον αφορά τους μεγάλους περιφερειακούς κινδύνους. Έδωσε σημασία σε αυτό. Και κυρίω οι πολλαπλέ μεταφορέ για τι στρατηγικέ που έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση κατά των πυρκαγιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα εκ μέρου των ε, μεταρρυθμιστών συντηρητικών, ο κύριος Βανέρσκι για 1,5 λεπτό. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo, Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, γιατί αποτελεί για μια, για μια ανάπτυξη 500% σε ό,τι αφορά την συχνότητα εμφάνιση φυσικών καταστροφών σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν αφορά, αφορά όμω μόνο το Πακιστάν, την ΑΕΤ, αλλά και την Ευρώπη, του Ευρωπαίου πολίτε που πέφτουν θύματα των καταστροφών αυτών. Και φυσικά υπόκειται και τις ε, υλικέ ζημίε. Είναι σημαντικό λοιπόν που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, γιατί είμαστε, αν είμαστε ειλικρινεί, τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κράτη-μέλη, δεν μπορούν πάντα να ανταποκριθούν σε αυτές τις καταστροφές. Αυτό αφορά και τη δική μου χώρα, την Πολωνία, όπου η κυβέρνηση απέτυχε και έχω υπόψη μου τα θύματα της τελευταίας φυσικής καταστροφής. Υπήρξαν πολλά θύματα που έχασαν όλο τους το βιός και τις επιχειρήσεις τους σε πολλές περιπτώσεις. Τα θύματα, ξέρετε, πρέπει να βοηθηθούν υλικά. Δεν ε, τους αρκούν τα σύμβολα. Όχι. Θέλουν υλική βοήθεια. Και είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να μην μιλάμε μόνο για την βοήθεια ex post, αλλά και για τη διάσταση της πρόληψης μιλάμε για τις πυρκαγιές, αλλά στην περίπτωση της Πολωνίας μιλάμε και για τις πλημμύρες. Και κυρία Πρόεδρε, τρίστε και το χρόνο. Το χρόνο. Ε, στον κατάλογό μου έχω επόμενο μιλητή τον κύριο Τρεμόπουλο, εκ μέρους των Πρασίνων, αλλά δεν είναι ακόμα στην αίθουσα. Έτσι θα περάσω στην κυρία Ντεμπράν, εκ μέρους της ε, Ενωτικής Αριστεράς. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά.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 όταν αυτές συμβαίνουν, είναι πολύ βασικό να βασιστούμε στους πυλώνες εκείνους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις φυσικές καταστροφές. Ο συντονισμός είναι ένα στοιχείο κλειδί αν θέλουμε αποτελεσματικά να προσφέρουμε την βοήθειά μας στον κόσμο. Συγχρόνως πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ανθρωπιστικές αρχές που έχουν να κάνουν με την αμεροληψία, με την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι, ανθρωπιστικές, οι ανθρωπιστικοί κανόνες θα ισχύουν. Οι καταστροφές δεν μπορεί ποτέ και αντιμετώπιση τους να έχουν να κάνουν με πολιτικούς παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια λοιπόν πρέπει να προσφέρεται ανεξάρτητα από πολιτικές ρυθμίσεις ή από πολιτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν την ανθρωπιστική αρρωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεμπρά. Τώρα ε, επόμενος ομιλητής ο κύριος Ρώση από την ομάδα Ελευθερίας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όπως και άλλοι την εισηγήτρια την κυρία Γκαρντίνη διότι κατάφερε να κάνει έξοχη δουλειά, είναι σαφές και όλοι γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις καταστροφών, φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών το καλύτερο θα ήταν να προληφθούν. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό κάτι τέτοιο. Παρ' αυτά όταν αυτές συμβαίνουν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να παρέμβουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον ταχύτερο δυνατό, στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Η συνθήκη τη Σαββόνα επιτρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί και στον τομέα τη προστασία των πολιτών. Άρα θα ήταν σκόπιμο σε περίπτωση καταστροφών είμαστε θέση να δημιουργήσουμε κέντρα διαχείριση των κρίσεων που θα είναι λειτουργικά 24 ώρε 24, 7 μέρε στι 7 θα πρέπει να αποφύγουμε την επικάλυψη του πολλαπλασιασμού των παρεμβάσεων και σε πολιτικό επίπεδο και λειτουργικό και επιχειρησιακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο πνεύμα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ανάγκη δεν θα πρέπει να υπάρχουν φραγμοί. Θα πρέπει να καταφέρνουμε να παρεμβαίνουμε γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Και μετά, εάν καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος στη στιγμή κρίσης, προφανώς δεν θα κάνει κακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόντερ Μάγερ τώρα για 1,5 λεπτό εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αντίδραση των καταστροφών, αλλά θα πρέπει να διδαχτούμε και από τις πρόσφατες καταστροφές προκειμένου τις ε, επικίνδυνες ε, τεχνολογίες όπως η ατομική ενέργεια να τις αποφύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν όλα αυτά και αυτά δεν έγιναν τα απαραίτητα, για παράδειγμα, στην προσφατή καταστροφή με την Λάσπη στην Ουγγαρία σε κάποιους τομείς ε, θεωρούμε ότι η αρχή της, ε, αυτό, της πρόληψης αυτής είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι κίνδυνοι αυτοί να αντιμετωπιστούν από τα κράτη-μέλη, όπως η Αυστρία για παράδειγμα, στο νότιο Τυρόλο. Η προληπτική αντιμετώπιση των καταστροφών είναι κάτι που υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τρεμόπουλος καθυστερημένα θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό εκ μέρους της, ε, της ομάδας των Πρασίνων. 1,5 λεπτό κύριε συνάδελφε αξιότιμοι συνάδελφοι θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη σύνταξη αυτής της ε, συνενετικής έκθεσης μιας έκθεσης που υπογραμμίζει ε, την ε, ανάγκη να αναβαθμιστούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί αντιμετώπισης των καταστροφών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που τόσο ανάγκη έχουμε αυτόν τον καιρό με τον ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό και ένταση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών ε, αυξάνει και η ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής διαχείρισης των καταστροφών συμπεριλαμβανομένων και της πρόληψης της ετοιμότητας αντιμετώπισης και της αποκατάστασης. στο λίγο χρόνο θα ήθελα να επικεντρωθώ στην πτυχή της πρόληψης. θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε χρήματα και χρόνο αν επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη παρά στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση ο αυξανόμενος ρυθμός της αλλαγής του κλίματος και η εξάντληση των φυσικών πόρων θα αυξήσει περαιτέρω τις πιθανότητες για συχνότερες και πιο έντονες φυσικές καταστροφές. η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων είναι μια έξυπνη προληπτική επένδυση που εκτός από ανθρώπινες ζωές θα σώσει και πολύτιμο πόρους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. σε αυτό το πλαίσιο οι τροπολογίε μας που υιοθετήθηκαν στην επιτροπή περιβάλλοντος τόνισαν ακριβώς αυτή τη διαπίστωση αλλά και την ανάγκη για πιο αποτελεσματική το σχεδιασμό απόκριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν πετρελαιοκυλίδε πυρηνικά και άλλα επικίνδυνα υλικά. τόνισαν επίση την ανάγκη να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά την αρχή ορυπαίνων πληρώνει όσο αφορά την ευθύνη για την περιβαλλοντική ζημιά. τα ε, ατυχήματα του κόλπου του μεξικού και τη φουκουσίμα δεν πρέπει να σβηστούν ποτέ από τη συνείδησή μα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλε, αν και ξεπεράσατε το χρόνο. Ερχόμαστε τώρα στον κατάλογο των επόμενων ομιλητών. Ε, έχει το λόγο ο κύριος Λάρντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νόμιζα ότι είχατε βγάλει από τη λίστα, αλλά πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Μου δίνετε το λόγο. καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Καρτίνη, η οποία νομίζω ότι ε, κατάφερε να φτιάξει μια έκθεση συνοπτική και σύντομη, η οποία όμω ε, είναι αξιοσημείωτη. Βλέπουμε ότι γίνεται αναφορά στις ε, νομικές βάσεις επί των οποίων βασιζόταν ως τώρα η δουλειά μας. Και νομίζω ότι τα τελευταία αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των καταστροφών καταδεικνύουν ότι α, ανταποκριθήκαμε σωστά. Αλλά αλλάζει και η κατάσταση στην Ευρώπη. Έχουμε όλο και πιο πολλές καταστροφές από πλευρά περιβαλλοντικών καταστροφών αλλά και τρομοκρατικέ επιθέσει. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομοθεσία. Θα προτείνει σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει να έχουμε το εξή ωστόσο υπόψη. Και αυτό το ακούσαμε διάφορες, σε διάφορε περιπτώσει. Ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αν θέλουμε ωστόσο μια υπηρεσία συντονιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι μπορεί να προκύψει μόνο από την ουσία των κρατών μελών. Αλλά ο συντονισμό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε πού βρίσκονται διάφορε υπηρεσίε, τι ικανότητα έχουν και να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον συντονισμό. Νομίζω ότι υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά πολύ σημαντικότερο θα είναι να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, η οποία είναι απαραίτητα. Κάτι άλλο τώρα για το Ταμείο Αντιμετώπισης Καταστροφών. Μιλάτε για ε, επέκταση αυτού. Εγώ είμαι κατά. Έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες ε, για την ε, χρησιμοποίηση του Ταμείου Καταστροφών που πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτές για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστροφών. Έτσι θα πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Στρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι φυσικές καταστροφές είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε ξανά και ξανά στο Κοινοβούλιο και διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο και πιο συχνά και όλο και πιο καταστροφικές τέτοιες φυσικές καταστροφές. Γι' αυτό και χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Επιτρόπου Γιώργεβα, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλή, πολύ σωστή και θέλω να συγχαρώ και την συγκίτρια, βέβαια, την κυρία Γκαρδίνη. Εμείς οι σοσιαλιστές συμφωνούμε με την ανάλυση που γίνεται όσον αφορά τα αίτια, τις κλιματικές αλλαγές, από τις οποίες απορρέουν όλο και περισσότερες και πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε τις πολιτικές μας πρόληψεις. Προβλέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρόπους για να ενισχύεται η αντίδρασή μας σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Πρέπει να είναι πιο συντονισμένη δηλαδή η αντίδρασή μας και πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό και μας ικανοποιεί η ιδέα να υπάρξει μια ευρωπαϊκή δύναμη αντίδρασης έκτακτων καταστάσεων. Πρέπει τα κράτη-μέλη να δώσουν πόρους, έτσι θα έχουμε και το Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Χάρη σε ένα σύστημα λειτουργικό που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και που θα λειτουργεί καλά διαρθρωμένο με τα κράτη-μέλη μέσα από κεντρικά σημεία, τα οποία επίσης θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις που κάνει όσον αφορά τα πειραματικά προγράμματα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πειραματικό πρόγραμμα για να υπάρξει ένα απόθεμα ε, αεροσκαφών έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δασικές πυρκαγιές. Πρέπει όντω να υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Η συνθήκη τη Λισαβόνα επίση. Μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ρήτρα αλληλεγγύη. Δημιουργεί αυτή τη ρήτρα αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράμε σε καταστροφέ. Γι' αυτό και εμεί θα έχουμε και τροπολογίε έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ιδέα τη αλληλεγγύη. Ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Παναγιώτοφ, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα και θα πάρει το λόγο ο κύριο Βλασάκ για 1,5 λεπτό. Ακριβώ 1,5 λεπτό, σα παρακαλώ, όχι παραπάνω. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι αν αντιμετωπιστεί σωστά η καταστροφή με δυνατότητα καλή αντίδρασης, μπορούν να σωθούν πολλές ζωές και τεράστιες καταστροφές μπορούν να αποφευχτούν. Η πρόληψη όμως φαίνεται ότι είναι η καλύτερη λύση από όλες. Κυρίως όσον αφορά τις ανθρωπογενείς καταστροφές όπως είναι η Φουκοσίμα, η καταστροφή του Μεξικού. Θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη ασφάλειας μέσω πρόβλεψης και πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή του κλίματος και την αναπτυσσόμενη οικονομία. Αν προσέξουμε σωστά, θα μπορούμε να μειώσουμε τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Θα ήθελα ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για τη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ σημαντικό αλλά πάρα πολύ περίπλοκο θέμα. Δύσκολο να βρεθούν κοινέ γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων που διαφέρουν το ένα από το άλλο. Και χρειάζεται πολύ ταχεία και ακριβής αντίδραση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Μπλουμ θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Well, I rise, uh, με κάποια ταπεινότητα μιλάω, εκπροσωπώντας μια χώρα που κατάφερε να εκλέξει Υπουργό Οικονομικών ε, Σκοτσέζο. Ο μόνος Σκοτσέζο που δεν ε, τον εννοιάζει πόσα χρήματα να ξοδεύσει. Μοναδικός. Λοιπόν, με κάποια ταπεινότητα μιλάω, έχοντα εκλέξει από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών. Όμως, προσβλέπω με το βρετανικό χιούμορ που διαθέτει το τα μεταφερέσει κανένα, Προσβλέπω πως αυτό το μέρος μας έδωσε ενεργειακή πολιτική, πολιτική απασχόληση, αλληλεία, γεωργική πολιτική. Σχεδόν τα πάντα που έκανε η Ένωση ήταν καταστροφή. Και τώρα θέλουμε να βρούμε μια αντιμετώπιση καταστροφής. Οι περισσότερε ανταποκρίσεις ε, δημιουργούνται εδώ, σε αυτό το χώρο. Δεν λέω ότι προσβλέπω να δω πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Και θα ήθελα να δω τι είδου τελικά χάλια θα καταφέρετε να κάνετε με αυτό το μέτρο. Κύριε Μπλουμ, η κυρία Γκροστέτ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συνάδελφος κυρία Καρδίνη εξήγησε πάρα πολύ καλά στην εισαγωγή της ότι πρόκειται για αλληλεγγύη, επικουρικότητα και αποτελεσματικότητα θα πρόσθετα εγώ, γιατί το είπαμε, οι φυσικές καταστροφές είναι όλο και περισσότερες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί. Είναι πολύ καλή η έκθεση που προηγουμένω ο Μισελ Μπαρνιέ είχε κάνει το 2006 και η έκθεση αυτή εμπνέεται από την έκθεση Μπαρνιέ, στην οποία έλεγε ο κύριο Μπαρνιέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τα μέσα που διαθέτει να τα βάλει από κοινού έτσι ώστε να δημιουργήσει κάποιο είδου ευρωπαϊκή μονάδα πολιτική προστασία να μπουν μαζί τα μέσα μας λοιπόν για να μπορούμε να αντιδράμε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Έχουμε και την τεχνολογία, έχουμε το πρόγραμμα Γαλιλαίο, έχουμε το πρόβλημα GMS, έχουμε επίσης τις τηλεπικοινωνίες. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε έγκαιρα, γρήγορα, ώστε να παρεμβαίνουμε και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και υπενθυμίζω όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες για παράδειγμα πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης κλήσης. Έτσι μπορούν να σωθούν χιλιάδες ζωές Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ζωτική σημασία οι πολίτες μας να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας αριθμός κλήσης για έκτακτη ανάγκη. Η έκθεση της κυρίας Γκαρδίνη δείχνει ότι μπορούμε όντως να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων χωρίς να αλλάξουμε τις υπάρχουσες δομές προσέχοντας να τηρείται πάντα επικουρικότητα, αλλά από την άλλη μεριά να βάζουμε από κοινού τα μέσα που διαθέτουμε γιατί αλλιώς κοστίζει περισσότερο η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Το συντονισμό αυτών πρέπει να τον φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι περιμένετε βοήθεια από το Κοινοβούλιο μας. Ε, λοιπόν, μπορείτε να βασιστείτε σε εμά για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Γκροστέτ. Τώρα ο κύριος Αρσένης θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό, κύριε Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε. Καταρχήν να συγχαρώ τους συναδέλφους που εργάστηκαν εντατικά για αυτή την έκθεση είναι μια έκθεση που από ό,τι φαίνεται και από τις ομιλίες των συναδέλφων υπήρξε μεγάλη και ευρία συνένεση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, ε, την κυρία Γκαρντίνη, αλλά και στον κύριο Σταυρακάκη από την Επιτροπή Περιφερειών. Είναι η δεύτερη έκθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα που ε, θα ψηφίσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έκθεση για την δασική προστασία που μας ζητά να πάρουμε μέτρα για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών τα ευρωπαϊκά δάση τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητα όμως για να προσαρμόσουμε προετοιμάσουμε τις κοινωνίες μας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. απειλούνται από την κλιματική αλλαγή ε, με πυρκαγιές ε, πλημμύρες και πάρα πολλά ακραία φαινόμενα όπως απειλείται όλη η ευρώπη με ακραία φαινόμενα ε, και αυτό μας υποχρεώνει είναι διασυνοριακά αυτά τα φαινόμενα και μας υποχρεώνει να πάρουμε μέτρα. απαιτείται και περιμένουμε την απάντηση της επιτροπής ε, για το αν θα προχωρήσει στη λευκή βίβλο για τη δασική προστασία αν θα έχουμε νομοθεσία για την προσαρμογή των δασών μας στην κλιματική αλλαγή και για δεύτερη φορά το κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή ζητά νομοθεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ένα μέτρο που εξοικονομεί πόρους και που είναι κρίσιμο σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Ε, όταν όμως συμβαίνουν οι πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα πρέπει να έχουμε έναν ευέλικτο μηχανισμό αλληλεγγύης προσαρμοσμένου στι τοπικέ ανάγκε που να μπορεί να απαντά, να έχει την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σένη, ήσασταν και συνεπή στον χρόνο. Ο, τώρα ο κύριος Γκέρεν θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν 36 διαφορετικοί τρόποι για να βελτιώσουμε την δυνατότητα αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι φυσικέ καταστροφέ. Χρειάζεται πρόληψη, συντονισμό, να βάζουμε από κοινού του πόρου μα. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Ε, πρόληψη ε, βασιζόμενη στην αηφόρα ανάπτυξη. Συντονισμό με την ανταλλαγή πληροφοριών επιμονήμου βάσεω. Και να βάζουμε από κοινού τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα κάνουμε και καλύτερη διαχείριση ε, του χρήματος των πολιτών μας. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, εμπόδια, πρέπει να έρθουν και τα τελευταία εμπόδια προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Γεωργέβα, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ακόμα σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά την τήρηση των αρχών αυτών και την επίτευξη κατά συνέπεια των στόχων που πρέπει να τηρήσουμε, το προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας εξάλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκουτιέρε, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή η έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη. Βέβαια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Θα ήθελα όμως πέρα από την πρόληψη να αναφερόμασταν και στην επόμενη μέρα. Γιατί ένα από τα κυριότερα προβλήματα που έχουμε στην Αϊτή ή στην Λόρκα της Ισπανίας μετά τον πρόσφατο σεισμό εκεί ή στην Άκουλα στην Ιταλία είναι ότι τι είναι επομένη, όταν δηλαδή σωθήκαν ό,τι ζωή σωθήκαν, μετά τους ξεχνάμε. Ενώ πρέπει να υπάρξει ανοικοδόμηση, να ξαναφτιαχτούν αυτές οι πόλεις και χρειάζονται πολλές φορές χρόνια για να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει επιστήμη, πρέπει να τους βοηθάμε. Δεν μπορεί μετά από ένα σεισμό να χτίσουμε οπουδήποτε. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία που μπορεί κανείς να χτίσει ή που δεν μπορεί να χτίσει. Άρα χρειάζονται τη βοήθεια αυτή, να βάλουμε τη γνώση που διαθέτουμε μαζί για να τους βοηθήσουμε. Λέμε ότι οι νέες ε, πόλεις θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικές, ενεργειακά κτλ. κτλ. Πώς θα το πετύχουμε όμως αυτό η Ευρώπη έχει εγκαταλείψει τελικά τους πολίτες της αυτούς. Δεν έχουν ε, λυθεί συντονιστικά μέτρα. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να συντονίσετε και την ανοικοδόμηση και να φροντίσετε για πραγματική πρόληψη. Στην περίπτωση των πλημμυρών γίνεται αυτό. Με τα ποτάμια. Η Ισπανία έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει πολλά, αλλού όχι. Δεν μπορεί λοιπόν την επόμενη μέρα να ξεχνάμε τη φυσική καταστροφή. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το τι γίνεται την επόμενη μέρα. Πάνω σε αυτό θέλω να δουλέψετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κουτιέρες. Η κυρία Χίμπνερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εξ ονόματος της ομάδας μας την ε, συνάδελφο Καρδίνη, η οποία προετοίμασε μια πάρα πολύ καλή έκθεση που περιλαμβάνει όλες τις αρχές και όλες τις προτεραιότητες που χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή ικανότητα αντίδραση και πρόληψης καταστροφών θα συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών και επιπλέον έχει να τριδραματίσει μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και έχω υπόψη μου ανθρωπιστικές ε, δράσεις σε χώρες που πλήττονται από τέτοιες φυσικές καταστροφές. Η πρόταση δημιουργίας Ευρωπαίων συμμάχων είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ελπίζουν να διατηρήσουν την πλήρη αυτονομία τους στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στους τομείς διάθεσης των πόρων τους και θα έχουν λοιπόν ε, τη δυνατότητα να διαθέτουν ανα πάσα στιγμή α, τις, τους πόρους αυτούς για την ευρωπαϊκή ελληνική. Πολλές ε, χώρες έχουν σχετικές υπηρεσίες για την ε, πρόληψη καταστροφών. Θα μπορούσαν λοιπόν να ανταλλάξουν σχετικές προτεραιότητες και σχετικές πρακτικές και αυτό θα βοηθούσε τον συντονισμό. Επίσης θα είναι σημαντικό να καταρτιστούν σενάρια για ενδεχόμενες μελλοντικέ φυσικές καταστροφές. Αυτό και για το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τις περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα κέντρο ε, και καταστροφών είναι και αυτό απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ε, Βεράκ τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια, όπω είπαν όλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επλήγει από καταστροφέ ανεπροηγουμένου και αν τι παραθέσουμε τι καταστροφές θα παίρνει όλο τον χρόνο. Έκρηση τη ε, ΑΖΕΝΤΕΦ πέρασαν 10 χρόνια στην Τουλούς το έγιναν, <laughs> θυμηθήκαμε αυτήν την επέτειο. Η έκθεση Yes είναι πραγματική δυνατότητα που μα δίνεται για να δείξουμε αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλληλεγγύη μεταξύ των λαών μα. Εδώ και αρκετά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει λειτουργική ε, την κοινή προσπάθεια και θα πρέπει όλοι μαζί να μπορούμε να κινηθούμε και να δράσουμε και να μην περιμένουμε μια νέα καταστροφή να πλήξει τις επικράτειές μας για να λύσουμε μαθήματα. Σήμερα θα πρέπει να διαθέσουμε στον καθένα τις υλικέ μας δυνατότητες και τις ανθρώπινες και τις οικονομικές για να αποφύγουμε νέα δράματα. Ε, κυρία Επίτροπε, είπατε προηγουμένω ότι θα πρέπει να προβλέπουμε τους κινδύνους. Και είναι πραγματικά λυπηρό ότι σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποσυρθεί από την χρηματοδότηση ε, του προγράμματος επιτήρησης και παρακολούθησης που θεωρείται από όλους ότι είναι ένα μέσο πάρα πολύ ουσιώδες για την πρόληψη και το συντονισμό ε, των απαντήσεων που τις καταστροφές. Και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της και να υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό που είναι φάρος και δίνει αναμφισβήτητη ε, υπεραξία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ την κυρία Γκαρντίνη για την πάρα πολύ καλή καλή έκθεση. Ελπίζω ότι θα την εγκρίνουμε, θα ανοίξει έτσι το δρόμο προς μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Ε, θα, δεν θα μπορέσουν να το πάρουν όλοι. Θα πάρουν το λόγο τρεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ένας από την αριστερά συνάδελφος που έχει ζητήσει και τρεις από την ομάδα των σοσιαλιστών παρόλο που έχουν ζητήσει περισσότεροι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Σκούρια. Ένα λεπτό παρακαλώ, δεν θα το ξεπερνάτε για να μπορέσουν να μιλήσουν οι συνάδελφοι που είπα. Ένα λεπτό κύριε Σκούρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη στιγμή, στο λεπτό που έχω στη διαθεσή μου, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη συνάδελφο την κυρία Καρτίνη για την έξοχη έκθεσή τη και διότι ε, με τι επαφέ που υπήρχαν με του διάφορου ε, φορεί καταλήξαμε αυτό το κείμενο. Χρειαζόμαστε περισσότερα. Θα πρέπει να έχουμε νομοθετικό ψήφισμα που να μπορεί να κάνει, είναι ένα βήμα προόδου και να διοργανώνει η προστασία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρί κενά και χωρί αλληλεπικαλύψει. Τη στιγμή που συζητεί το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτό είναι το πλαίσιο εντό του οποίου υπάρχει απέτηση για περισσότερη Ευρώπη για να δώσουμε ζωή σε μια ενωτική και συντονισμένη δράση σε όλη την Ένωσή μα κυρίω διότι η προστασία των πολιτών ζει από την ελληνική και την εθελοντική δράση που εντάσσεται ε, και στην συνθήκη της Αβώνας και στο ευρωπαϊκό έτος της εθελοντικής προσφοράς. Και ε, χρειάζεται και μια οικονομική επένδυση. Γι' αυτό ευχαριστώ την Επίτροπο που το υπογράμμισε αυτό σαν πτυχή και ζητώ αύξηση των κονδύλιων. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Σκούρια. Η κυρία θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ταμείο Ελληνικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως λειτουργεί καλά, αλλά τον πρώτο χρόνο που το εφαρμόσαμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και περιορισμοί και αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την έλλειψη άμεσης αντίδρασης κάθε φορά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά και κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή κριτήρια ή επειδή δεν ορίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και καλά το ότι είναι φυσική καταστροφή. Ευτυχώς τώρα έχουμε κάποια προγράμματα. Πάντως η χρήση των κονδυλίων αυτών έχει διαπιστώθει ως προβληματική. Γι' αυτό και πιστεύω πως η δυνατότητα προσφοράς αρρωγής που να βασίζεται σε μια αρχική εκτίμηση σε μια χώρα που πλήττεται από φυσική καταστροφή είναι κάτι που θα μας διευκολύνει πολύ μετά από μια καταστροφή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα θα πάρει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ. Πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2010, η μεγάλη πλειονότητα και η μεγάλη πλειοψηφία εδώ του Κοινοβουλίου ε, ενέκρινε τη δική μου έκθεση για μια κοινωτική αντίδραση σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Συζητήσαμε το θέμα της πρόληψης και το πώς θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διάσταση αυτή. Η πρόληψη μπορεί πραγματικά να σταματήσει πολλές ε, καταστροφές και να απαλύνει την έκταση άλλων. Στην έκθεση αυτή συζητήσαμε και το κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο για την πρόληψη, για την προστασία των δασών, των ακτών, των ε, υδροφόρων οριζόντων ένα σύστημα ελάχιστη αποζημίωσης για τους αγρότες που πλήττονται από καταστροφέ και για ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίηση. Ένα χρόνο αργότερα τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πολύ στάσιμα. Τι κάνουμε, μιλάμε μόνο για τη συνεργασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πράξουμε και όχι να μιλάμε. Πρόεδρε, να μην ξεπεράσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχουμε μία παροιμία που λέει ότι οι καταστροφές πλήττουν τους ανθρώπους και όχι τα βουνά. Είναι λοιπόν ουσιώδες να χορηγείται βοήθεια αρρωγή. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να καλωσορίσουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτόνομου κέντρου αντίδρασης σε τέτοιες καταστροφές για την παροχή της ανθρωπαστικής βοήθεια και την χορήγηση, την ε, συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας σε υλικό επίπεδο, αλλά και πιστεύω ότι με, την... τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ζωή των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επί αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση του αριθμού των καταστροφών, ανησυχητική αύξηση και γίνονται όλο και πιο σοβαρές οι καταστροφές. Οι καταστροφές που πλήττουν τα κράτη-μέλη και τα κράτη σε όλο τον κόσμο, ε, μα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένα φορέα που θα τη δρά γρήγορε καταστροφέ. Και τα γεγονότα που οδηγούν στι καταστροφέ δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά μπορούμε να τα χειριστούμε. Ο κίνδυνο που σχετίζεται με τα φυσικά φαινόμενα θα πρέπει να μειώνεται μέσω μέτρων. Μέτρων πρόληψη, για να μειώνεται η συνέπεια τη καταστροφή οικονομική ενίσχυση πάνω από 200 δις ευρώ που δόθηκε κατά την περίοδο 2008-2010 από το Ταμείο Αλληλεγγύης αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βοηθήσει. Όμως τα χρήματα δεν φτάνουν εύκολα σε εκείνους που έχουν πληγία τις καταστροφές. Χρειάζεται ένας μηχανισμός λοιπόν που θα βοηθά το χρήμα να φτάνει πιο γρήγορα στον κόσμο που πλήττεται. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταμπάτσι θα πάρει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Λέει στα ελληνικά ο μιλητής. Τις καταστροφές τις έχει γνωρίσει και η Ουγγαρία πολύ πρόσφατα μετά από μια βιομηχανική καταστροφή. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθησε πολύ την Ουγγαρία, πράγματι εποφεληθήκαμε από την βοήθεια αυτή. Διαπιστώσαμε όμως ότι ήταν μια χειρονομία ad hoc, δηλαδή μια πρωτοβουλία σαν και αυτή που έχουμε στη σημερινή έκθεση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να εκφράσω όλες τις ευχαριστίες μου επίσης στην Επίτροπο, αλλά και στο σύνολο του ημικυκλίου εδώ. Γιατί πραγματικά πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε πολύ καλά το όνομα της κυρίας Γεώργιεβα, γιατί έχει βοηθήσει πολύ. Θα σας ε, μιλήσω τώρα και για κάτι άλλο, για την παρέμβαση των αρχών. Για τόσα επιβάλλονται στην περίπτωση της Ουγγαρίας, οι καταστροφές είναι έξι φορές παραπάνω από την αξία της επιχείρησης που την προκάλεσε. Η κυρία Λούκα Σιέμφσκα έχει το λόγο τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, δεδομένων ε, δεδομένη τη συχνότητα των καταστροφών, θα πρέπει όντω να αντιδράσουμε γρήγορα και συντονισμένα και με το βέλτιστο τρόπο να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να περιορίσουμε τις ίλικές ζημίες. Και χαίρομαι που σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη και στην έκθεσή σας οι σχετικές οργανώσεις. Αυτές αποτελούν άλλωστε την πρώτη γραμμή στην καταπολέμηση και τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών. Επίσης χαίρομαι για την πιο ευέλικτη διαμόρφωση του Ταμείου Αλληλεγγύης, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτοί που έχουν πληχθεί από καταστροφές επί σειρά εβδομάδων, μηνών να περιμένουν τη βοήθεια, την ε, ηλικία αυτή βοήθεια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ελπίζω όλα τα στοιχεία της έκθεσης να εφαρμοστούν, να βελτιωθεί η αντίδραση. Ο πολλαπλασιασμός των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών είναι γεγονό και ταυτόχρονα τα εθνικά μέσα που είναι διαθέσιμα για ανταπόκριση είναι όλο και λιγότερα και βρίσκονται υπό ένταση διότι ο κόσμος περιμένει βοήθεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα ήταν ανταπόκριση και ad hoc και γραφειοκρατική. Χρειάζεται γενική αναδιάθρωση του συστήματος. Και η λεπτομερέστατη αυτή έκθεση παρέχει του αναγκαίου προσανατολισμούς. Πρέπει να εξαλείψουμε τις επικαλύψεις και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των μέσων που διαθέτουμε. Πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την πρόληψη από την αντίδραση. Χρειάζεται εποπτεία, προετοιμασία, εκπαίδευση. Χρειάζεται μόνιμη διοργάνωση των εθνικών μέσων που θα διατίθεται για σκοπούς. Αύξηση ευελιξίας των διαδικασιών, ώστε το σύστημα να γίνει πιο λειτουργικό και θα πρέπει να επικρατεί η επικουρικότητα, να διατίθεται τα μέσα και τα χρήματα. Η προστασία των πολιτών πρέπει να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της παρέμβασης, τονίζεται το πολιτικό στοιχείο έναν του στρατιωτικού, που ακόμα και αν δεν εξαλείφεται εντελώς δεν θα είναι στο και επίκεντρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα τελευταία παρεμβαίνουσα η κυρία Κώστα για ένα λεπτό, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη και την ε, Επίτροπο και θέλω να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη χρειάζεται νομοθεσία ευρωπαϊκή, χρειάζεται εκ των κάτω προ τα άνω προσέγγιση, χρειάζεται καλύτερη, καλύτερο συντονισμό που θα συντονίζει τι εμπειρίε και τα μοντέλα παρέμβαση για την προστασία των πολιτών των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνουν εθελοντική παρουσία, εθνικό συντονισμό, συμμετοχή των τοπικών φορέων. Η ενίσχυση του 112 πρέπει να είναι ενιαίο ε, νούμερο κλήση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ γι' αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια παλήθευση, να δει στη χώρα μου Κινόμαστε προ κατακαιρματισμό των αριθμών που χρησιμοποιούνται και των δομών ανταπόκριση στι επίγουσες κλήσει. Δύο αριθμοί υπάρχουν για τι πυρκαγιέ, παραδείγματο χάρη. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στις τεχνολογίε μα όσον αφορά το pre-warning και το warning, υποστηρίζοντα την εφαρμογή των διαφόρων ε, μέσων που δεν χρηματοδοτούνται παρκούς. Χρειάζεται διοργάνωση προστασία των πολιτών και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πάνω σε αυτό τι κοινωνικέ αλλαγέ που χρειάζονται και που έγιναν όσον αφορά την Ευρώπη. Ε, ε, θα πρέπει, έχουμε περιφερειακές υποδομές αποκεντρωμένες. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούμε να ε, υποστηρίζουμε και τους πιο εύθραστους ε, πληθυσμούς. Κυρία Επίτροπος, Mrs. Commissioner, the floor is yours. Thank you. Ευχαριστώ πολύ για τα εξαιρετικά σχόλια και τις προτάσεις που άκουσα για την νομοθετική πρόταση. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις απαντήσεις μου ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με το τι θα κάνει η πρόταση αυτή που προσπαθεί να βάλει από κοινού τις δυνατότητες που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Η κυρία Στίφλε πρώτα απ' όλα το έθεσε αυτό. Είχαμε και μια σχετική ερώτηση από την κυρία Κροστέτ που λέει ποια είναι η σχέση όλων αυτών με την έκθεση Μπαρνιέ. Τι προτείνουμε εμείς λοιπόν. Εμείς προτείνουμε να βάλουμε μαζί τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Πρόκειται δηλαδή περισσότερο ε, από ό,τι έκανε ο κύριος Μπαρνιέ. Στην έκθεση Μπαρνιέ βλέπετε όπου έχουμε υιοθετήσει 12 προτάσεις ήδη, η ιδέα ήταν να βάλουμε από μαζί να βάλουμε μαζί τι δυνατότητε των κρατών μελών, αλλά η προσέγγιση ήταν περισσότερο από πάνω προ τα κάτω. Ενώ αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε τώρα είναι το αντίθετο, από κάτω προ τα πάνω. Και μπορώ να σα πω με σιγουριά ότι έχουμε τη στήριξη των κρατών μελών για την πρόταση αυτή, ιδιαίτερα από τι χώρε μέλη όπου. Σε εθνικό επίπεδο αυτό που θέλουν είναι να μην λαμβάνονται αποφάσεις μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, αλλά και σε πιο χαμηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν, έτσι μπορούμε να έχουμε μια δύναμη, θα έλεγα, στην οποία συγκεντρώνονται οι δυνατότητε των κρατών μελών. Και θα έλεγα μάλιστα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική πρόταση και δεν την περιμένουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχουμε ήδη βάλει μαζί τις δυνατότητες των κρατών μελών. Όταν εγώ ανέλαβα, είχαμε λιγότερο από 40 modules το οποίο είχαν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας πω ότι έχουμε 120 σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη, συν 8 συντονιστικές ομάδες. Έτσι λοιπόν προχωράμε για να ανταποκριθούμε ακριβώς στις ανάγκες. Και μάλιστα προς ενημέρωσή σας, το 2010 δραστηριοποίησαμε τον μηχανισμό άμεσης αντίδρασης 28 φορές. Τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή μπορεί να ήταν 2, 3, άντε 5 φορές. Ενώ αυτή τη φορά ήδη 11 και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις όπου θα δραστηριοποιηθεί ο μηχανισμός αυτός. Κάτι άλλο το οποίο έθιξαν πολλοί ευρωβουλευτές εδώ σήμερα, ο κύριος Αρσένης για παράδειγμα, ο κύριος Ζαλνέσκι και συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά του, η κυρία Ντεμπριν και άλλοι, είναι το εξή. Είναι η σημασία που έχει πρόληψη και η αποκατάσταση. Ξέρουμε ότι ένα ευρώ το οποίο ε, δίνουμε, επενδύουμε στην πρόληψη, είναι σαν να δίνουμε 4 ή 7 ευρώ στην αποκατάσταση. Παρ' όλα αυτά ήταν δύσκολο μέχρι τώρα και στην Ευρώπη αλλά και αλλού στον κόσμο να κάνουμε την πρόληψη αυτή. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Επιστρέφω από την Ουάσιγκτον μόλις, όπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγηθήκαμε με την Παγκόσμια Τράπεζα και με την κυβέρνηση της Ιαπωνίας για να θέσουμε το θέμα αυτό της ε, πρόληψης και της προετοιμασίας και να το βάλουμε ως πρώτη προτεραιότητα. Και θα συνεχίσουμε με διαρθρωτικά μέτρα που θα επικεντρώνονται σε ε, δραστηριότητες υπέρ της πρόληψης. Θα επανέλθουμε με μια επιπλέον νομοθετική πρόταση επ' αυτού όσο προχωράμε ε, στο λειτουργικό σκέλος. Βέβαια, οι δασικές πυρκαγιές φυσικά και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και όντως έχουν να κάνουν ε, οι καταστροφές των δασών με τις πλημμύρες, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές, γιατί και για το οικολογικό μας σύστημα έχουν μεγάλη σημασία και για τους πολίτες μας. Οπότε οι δασικές πυρκαγιές έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο δικό μας το έργο, κύριε Σένη. Η προετοιμασία βέβαια σημαίνει και από κοινού κατάρτιση. Και εδώ είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προωθήσει τον ρόλο μας. Την Παρασκευή που μας πέρασε ήμουν στην Πολωνία και εκεί συμμετείχα σε μία άσκηση προετοιμασίας πέντε χωρών. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι βάζοντας μαζί την πολιτική μας προστασία από κοινού είναι μια προϋπόθεση για να σώζουμε ζωές και για να χρησιμοποιούμε καλά τις δυνατότητες που έχουμε. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να κάνει περισσότερα σε αυτό το τομέα. Τώρα, κύριοι Λίνεν και Σίμπερ, είπαν πώς συντονιζόμαστε με την το εκπρόσωπο. Εδώ μπορώ να σας απαντήσω πολύ θετικά, ότι δηλαδή βάσει των ε, δράσεών μας σε περιπτώσεις κρίσης έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ την θεσμική συνεννόηση και τα πράγματα είναι πιο ξεκαθαρά τώρα για το ποιος κάνει τι, που και πότε. Και για να σας το διαρθρώσω αυτό ακόμα καλύτερα, μέσα στην Ευρώπη η ύπατη εκπρόσωπος δεν έχει ρόλο. Τα δύο τρίτα των παρεμβάσεών μας την προηγούμενη χρονιά ήταν μέσα στην Ευρώπη. Οπότε είναι θέμα εσωτερικής ευρωπαϊκής δράσης. Τώρα εκτός Ευρώπης εμείς δρούμε ως πρώτος αντιδρών ε, προσφέροντας πολιτική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια. Ενώ η ύπατη εκπρόσωπος έχει έναν πολιτικό ρόλο όπως επίση και στην άμυνα. Βέβαια σε περίπλοκες κρίσεις η ύπατη εκπρόσωπος αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και εμεί βοηθάμε με τις δικές μας δυνατότητες. Αυτή είναι η βέλτιστη πρακτική και στα κράτη-μέλη όπου η πολιτική προστασία συντονίζει και τα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά έχουν όπως ξέρετε τα δικά του κέντρα συντονισμού. Από την άλλη μεριά υπάρχει η πολιτική και η άμυνα που άλλοτε δεν έχει καθόλου ρόλο, άλλοτε συμμετέχει, εξαρτάται από την κρίση. Εσείς που είδατε τον πρόεδρο Ομπάμα να απαντάει ε, στις ε, πλημμύρες πρόσφατα, το έκανε από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Από την άλλη μεριά όμως, όταν έχει να κάνει με την περίπτωση του Μπιν Λάντεν, τότε ήτανε στο Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στο Λευκό Οίκο. Άρα είναι διαφορετική η ρόλη μας, αλλά φυσικά και πρέπει να συντονιζόμαστε μεταξύ μας σε ε, περίπτωση έκτακτων περιστάσεων. Και ανάλογα με τις έκτακτες περιστάσεις ε, οργανώνουμε και αποφασίζουμε για το πώς θα δράσουμε. Τώρα, τι εμπόδια υπάρχουν στα κράτη-μέλη, με ρωτήσατε. Το βασικό είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να καταλαβαίνουν ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά και σεβόμαστε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι η πολιτική προστασία οργανώνεται από τα κράτη-μέλη. Το σεβόμαστε αυτό, όπως επίσης και το γεγονός ότι σε εθνικές καταστροφές, όταν δεν υπάρχει ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δηλαδή η χώρα μέλος μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα, εννοείται ότι δεν θα παρέμβουμε. Και βέβαια τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε δύσκολες δημοσιονομικές καταστάσεις θέλουν να ξέρουν ότι εμείς θα φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Και εδώ απαντάω ότι ναι, θα φροντίσουμε κάθε ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου να δαπανηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Δηλαδή σε κοινοτικό επίπεδο όταν αυτό έχει νόημα, σε επίπεδο χώρας. μέλος όταν εκεί έχει περισσότερο νόημα. Με ρωτήσατε επίσης τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Είναι ένα ζωτική σημασία θέμα αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε και για την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Η αρρωγή για την ανάπτυξη με ε, τεχνικά μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να έχει στη διάθεσή της κάθε χώρα η οποία πλήττεται από φυσικές καταστροφές. Και έχουμε ήδη πάρει σχετικά μέτρα προκειμένου να βελτιώσουμε την αντίδρασή μας και την αξιολόγησή μας μετά από μια φυσική καταστροφή και να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή αρρωγή να συντονιστεί αντίστοιχα. Πάντως, συμφωνώ μαζί σας για το ότι αυτός είναι ένας τομέας πάνω στον οποίο πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Και είναι προτεραιότητά μας με τον συνάδελφο Πίβελς για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνώ επίσης με την κυρία Ντεμπρέν για το ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας κάθε φορά που παρεμβαίνουμε με ανθρωπιστική αρρωγή και με πολιτική προστασία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ιδιαίτερα σε σημεία που έχουν να κάνουν και πλήττονται όχι μόνο από φυσικές καταστροφές αλλά και από συγκρούσεις επιτόπου. Τις αρχές αυτές τις στηρούμε πάντα. Και ευχαριστώ και την ε, Βαρόνι Άστον που έχει βοηθήσει και εκείνη να τηρείται αυτή η αρχή της ουδετερότητας. Άλλοι ομιλητέ τώρα. Η κυρία Νταντσίλα, για παράδειγμα, είπε κάτι και πάλι συγγνώμη αν προφέρω άσχημα το όνομα, αναφέρθηκε στο Ταμείο Λιλεγγύης. Με τον Επίτροπο Χάν θέλουμε να υποβάλουμε πρόταση προκειμένου να επανορίσουμε το Ταμείο αυτό και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μια προχρηματοδότηση, μια προκαταβολή για χώρες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Όταν στην Μολδαβία και στη Ρουμανία είχαμε πλημμύρες, στη Μολδαβία μπορούσαμε να δώσουμε κοινοτική αρρωγή εν μία νυχτή, ενώ στην Ρουμανία όχι. Και γι' αυτό θέλω και εγώ να φροντίσω ώστε η αλληλεγγύη να προσφέρεται τη στιγμή που τη χρειάζεται ο κόσμος, τη στιγμή της φυσικής καταστροφής. Όσο και το Τζίμες είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι στον κατάλογο προτεραιοτήτων όσον αφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στηρίξει και οικονομικά το Τζίμις όσο γίνεται περισσότερο ε, με τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές, το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και εννοείται ότι θέλουμε και το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει. Και τέλος, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, όσον αφορά το αποθεματικό για την καταπολέμηση πυρκαγιών, εδώ τελειώνει, τελειώνει βέβαια τα κονδύλια του ταμείου το ταμείο αυτό ολοκληρώνεται δηλαδή και πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική πρόταση. Εδώ όμως δυσκολευτήκαμε με τα κράτη-μέλη, γιατί κάποιες χώρες μας δεν το θέλουν. Οπότε χρειαζόμαστε τη δικιά σας στήριξη. Όντως πρέπει να γίνει, το έχουμε δει ότι χρειάζεται, αλλά πρέπει ακόμα να δουλέψουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη για το ότι αυτή, αυτός ο δημοσιονομικός ε, διακανονισμός ε, χρειάζεται και πρέπει να συνεχιστεί. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά υπήρχαν πολλές και καλές ερωτήσεις και δεν ήθελα να αφήσω καμία απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Τώρα η συγγήτρια κυρία Γκαρντίνη για ένα μόνο λεπτό, διότι είχε περισσότερο χρόνο στην πρωτολογία της. Ένα λεπτό κυρία Γκαρντίνη, θα κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ήδη είχα υπολογίσει να αντικαταστήσω αυτά που μου κλάπηκα στην αρχή. Ένα λεπτό έχω. Δεν έχω να προσθέσω κατά τα λοιπά πολλά, διότι νομίζω ότι εδώ στη συζήτηση στην Ολομέλεια επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα, μεγάλη δυνατότητα που έχουμε σε αυτή τη φάση να είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι και να δώσουμε περισσότερη Ευρώπη στους πολίτες μας, να δώσουμε μια Ευρώπη που πολλές φορές δυστυχώς ήταν απόμακρη. Αυτή τη φορά όμως έχουμε ένα μέσο εξαιρετικό για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε μέσω Ευρώπη στον κόσμο με μικρά πράγματα, πέρα από τα βασικά θέματα που δεν πρέπει να τα επαναλάβω τώρα, δηλαδή πράγματα που φαίνονται όπως είναι ο αριθμός, το 112, ο αριθμός κλήσης ή το άρθρο 23 των συνθήκων, όπου εκεί αναφέρει ότι θα πρέπει να γνωρίσουν οι, οι πολίτες να το μάθουν. Ένας Ευρωπαίος πολίτης που είναι σε τρίτη χώρα και όπου η χώρα γέννησης δεν εκπροσωπείται, πρέπει να προστατεύεται από οδήποτε διπλωματικό σώμα οδήποτε μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει αυτή την Ευρώπη, αυτή χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ και καλή δουλειά στην Επίτροπο κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Και έτσι κλείνει η συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12.30. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη περνάμε στο επόμενο σημείο, στην ε, έκθεση του κυρίου Κασπάρη για τη νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της